Ε, επίσης η Γκουε ζήτησε η κυρία Πάφθη χθε του κυρίου Μαστάλκα να είναι μέλος της ε, νομικής επιτροπής και το ΙΝΕΒ ζήτησε ο κύριος Κολομπιέ να ενταχθεί στην Επιτροπή Γεωργίας και της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Υπάρχουν ενστάσεις, όχι